Επανάληψη της Συνόδου. Θα ήθελα να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα του... της τρίτης ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα είναι τα εξή. Τελικές ψηφοφορίες. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναπηρία μετά το 2020 εγκρίνεται τροποποίηση κάποιων κανονισμών όσον αφορά τι προσαρμογέ για την αντιμετώπιση τη πανδημία. Εγκρίνεται. Πολιτική ανταγωνισμού. Εγκρίνεται. Υποεπιτροπή για φορολογικά θέματα. Εγκρίνεται. Σύσταση Ειδική Επιτροπή για την καταπολέμηση του καρκίνου. Εγκρίνεται. Σύσταση Ειδική Επιτροπή για τι εξωτερικέ παρεμβάσει. Εγκρίνεται. Σύσταση Ειδική Επιτροπή για την τεχνητή νοημο... νοημοσύνη. Εγκρίνεται. Ε, Αρχικό κείμενο, παράγραφος 11, ε, εγκρίνεται. 14, πρώτο τμήμα, εγκρίνεται. 14, δεύτερο τμήμα, εγκρίνεται. Παράγραφος 20, εγκρίνεται. Παράγραφος 21, εγκρίνεται. Παράγραφο 45, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα εγκρίνεται, τρίτο τμήμα εγκρίνεται Το ψηφίσματο για την Τσεχική Δημοκρατία. Παράγραφο 49. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Α σε δύο τμήμα. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα επίση εγκρίνεται. Έκθεση για τα Δυτικά Βαλκάνια. 32 τροπολογία απορρίπτεται. Τροπολογία 33 απορρίπτεται. Τροπολογία 34 απορρίπτεται. Τροπολογία 35 απορρίπτεται. Τροπολογία 9 εγκρίνεται. Τροπολογία 10 εγκρίνεται. Παράγραφος 1. Αρχικό κείμενο, σημείο S, εγκρίνεται. Τροπολογία 36, απορρίπτεται. Παράγραφος 1, σημείο τι εγκρίνεται. Τροπολογία 11, εγκρίνεται. Τροπολογία 12, εγκρίνεται. Τροπολογία 13, εγκρίνεται. Τροπολογία 37, απορρίπτεται. Παράγραφος 1, σημείο AQ, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα εγκρίνεται και τρίτο τμήμα επίσης εγκρίνεται. Τροπολογία 14 εγκρίνεται, τροπολογία 38 απορρίπτεται, τροπολογία 39 απορρίπτεται, τροπολογία 15 εγκρίνεται, τροπολογία 40 απορρίπτεται, τροπολογία 16 εγκρίνεται, τροπολογία 41 απορρίπτεται, τροπολογία 17 σε δύο τμήματα, το πρώτο τμήμα εγκρίνεται, και το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Τροπολογία 42 εγκρίνεται. Τροπολογία 18 εγκρίνεται. Τροπολογία 19 εγκρίνεται. Τροπολογία 20 εγκρίνεται. Τροπολογία 21 εγκρίνεται. Τροπολογία 22 εγκρίνεται. Τροπολογία 23 εγκρίνεται. Τροπολογία 24 εγκρίνεται, τροπολογία 1 εγκρίνεται, τροπολογία 2 εγκρίνεται, τροπολογία 3 εγκρίνεται, τροπολογία 4 εγκρίνεται, τροπολογία 25 απορρίπτεται, η τροπολογία 26 απορρίπτεται, η τροπολογία 27 επίση απορρίπτεται, η τροπολογία 5 εγκρίνεται, το, η σκέψη J εγκρίνεται, η τροπολογία 28 απορρίπτεται, η τροπολογία 6 εγκρίνεται, η τροπολογία 7 εγκρίνεται, η τροπολογία 8 εγκρίνεται, η τροπολογία 29 απορρίπτεται, η τροπολογία 30 απορρίπτεται, η τροπολογία 31 επίση απορρίπτεται. Τροπολογία 10 εγκρίνεται, τροπολογία 5 απορρίπτεται, τροπολογία 1 απορρίπτεται, τροπολογία 11 απορρίπτεται, τροπολογία 6 απορρίπτεται. Παράγραφος 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα επίσης εγκρίνεται. Τροπολογία 7 απορρίπτεται. Παράγραφος 17 αρχικό κείμενο εγκρίνεται. Τροπολογία 2 απορρίπτεται. Τροπολογία 3 απορρίπτεται. Παράγραφος 24. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται και το δεύτερο εγκρίνεται επίσης. Παράγραφος 26. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα επίση εγκρίνεται. Τροπολογία